Euh, Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά ε, έλαβε χώρα μια τριμερή διάσκεψη για το NDCI, οπότε καθυστερήσαμε λίγο. Ανιέσκα Λαμάρ, υπεύθυνη ε, για τις ε, δικαστικές και αυθέτες εκτελέσεις του ε, ειδική εισηγήτρια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών της ΥΠΑ Αρμοστίας του ΙΕ. Συναντήκαμε ήδη στην Νέα με την κυρία Καλαμάχ. Συζητήσαμε τα θέματα του αγώνα εναντίον της ατιμορρησίας. Ε, είστε υπέρ της δημιουργίας ενός ε, παρατηρητηρίου για την ατιμορρησία είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων εδώ. Έχετε κάνει μια έρευνα για το θάνατο του ε, δημοσιογράφου Τζαμαλ Κασόγκη. Στην έκθεσή σας αναφέρετε ότι ο θάνατός του ήταν ε, προμελετημένη δολοφονία ε, και την ευθύνη είχε το κράτος της Αραβίας. Επίσης έχετε πιστεί στην προσοχή μας στις Φιλιππίνες και στην ε, κατάσταση που επικρατεί εκεί λόγω της καταστολής εκ μέρους του Πρόεδρου Ροντρίγκο Ντουάρτε με χιλιάδες νεκρούς. Ε, πολλές εντολές του ΟΕΕ καλύπτουν τον αγώνα αντίον της ατιμορρησίας σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του διεθνού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, εδώ είμαστε πολύ, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να δούμε τι έγινε ε, με αυτές τις εντολές και να ακούσουμε και τις ε, συστάσεις σας για την ενίσχυση της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου ήρθαμε σε επαφή με πολλούς αγωνιστές ε, των, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλοι μας σχολιάζουν το θέμα της ατιμορρησίας, διότι πραγματικά δεν υφίσταται απονομή δικαιοσύνη αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα πρόσβαση ανοιχτή πρόσβαση στην δικαιοσύνη και οι κατάλληλε κυρώσει. Το βλέπουμε αυτό και στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα στην Αμαζονία. Μας ε, ενημέρωσαν για το πώς η ατιμορρησία ε, των εταιριών αλλά και της κυβέρνησης και των κρατικών αρχών οδηγεί σε καταχρήσεις ε, και σε παραβίαση των κανόνων και του δικαίου. Έχετε το λόγο, κυρία Καλαμάχ, για 10 λεπτά. De, Προφανώς μπορείτε να μιλήσετε στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Έχω ετοιμάσει την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη από τους γαλόφωνους φίλους μου και τους γαλόφιλους. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για την ατιμορρησία. Δεν θέλω να ξεπεράσω το χρόνο μου, οπότε θα εστιάσω σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, καταρχήν σε ό,τι αφορά την ατιμορρησία και μετά θα κάνω θα σας μιλήσω για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις οποίες έχω ασχοληθεί. Ε, θα εστιάσω στην ατιμορρυσία σε σχέση με ανθρωποκτονίες. Για δολοφονίες βασικά, αυθόρ, ε, αυθαίρετες δολοφονίες ε, και μαζικές δολοφονίες. Σε ό,τι αφορά την ατιμορρυσία, το πρώτο που μπορώ να πω είναι προφανές αυταπόδεικτο, αλλά πρέπει να το πούμε ότι η ατιμορρησία είναι κάτι το συστηματικό. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα σύστημα. Ε, μια δολοφονία είναι πάντοτε μια δολοφονία. Αυτά που ακολουθούν όμως απαιτούν την κινητοποίηση μια σειράς μηχανισμών. Και όταν τελικά η ε, επικρατήσει ατιμορρησία σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποτύχει. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που έχει αποτύχει. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η ατιμορρησία ως έννοια, διότι αποδεικνύει το πώς ε, ε, αποτυγχάνουν τα όργανά μας, οι μηχανισμοί μας. Η ατιμορρησία λοιπόν είναι ένα συστημικό ζήτημα. Δεύτερον, Στην μακρά μου καριέρα ως αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, αντελήφθη ότι ε, μπορεί να έχουμε κουρδίσει το κοινό ε, σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, τους λέμε ότι μπορούν να βρουν απάντηση τα προβλήματά τους μέσω της δικαιοσύνης. Όμως ελάχιστα από τα αδικήματα σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων ε, καταλήγουν σε, στα δικαστήρια. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση απογοήτευσης, μια αίσθηση αποτυχίας του εθνικού ή του διεθνούς δικαιοδοτικού συστήματος. Προφανώς δεν προτείνω επουδενή να προσποιηθούμε ότι η δικαιοσύνη δεν συνδέεται με την εκδίκαση. Όμως θα πρέπει να δώσουμε ένα πιο ευρύ νόημα στην έννοια της δικαιοσύνης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι δικαιώθηκαν ή ότι μπορούν να δικαιωθούν χωρίς απαραίτητα να περάσουν από ένα δικαστήριο και από μια ε, δικαστική απόφαση. Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν οι προσδοκίες των ανθρώπων και των θυμάτων και να τους δώσουμε διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση με την απονομή της Δυνατότητες που δεν θα περιορίζονται σε μια εκδίκαση δυνατότητες να αποζημιωθούν ηθικά και υλικά με άλλο τρόπο και να αισθανθούν ότι δικαιώθηκαν. Καταλαβαίνω ότι αυτό το μήνυμα είναι ε, περίπλοκο. Αλλά μιλώντας με θύματα σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότερο πείθομαι γι' αυτό. Ίσως να έχουμε υπερβάλει λέγοντας ότι η μόνη δυνατή δικαιοσύνη για κάποια συγκεκριμένα ε, αδικήματα ε, είναι ε, αυτά τα αδικήματα να γίνουν αναγνωριστούν από ένα δικαστήριο ως ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για παράδειγμα γενοκτονία. Νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει συνεισφέρει στη δημιουργία μιας τέτοιας εντύπωσης ε, και μιας τέτοιας νοοτροπίας και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε χτίσει υπερβολικές προσδοκίες για το ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ε, και το περιεχόμενο μάλλον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα αυτές τις προσδοκίες δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι, ε, έχει αργές διαδικασίες, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, πολλούς παράγοντες, εγγυήσει, διαδικασίες. Πρέπει η δίκη να είναι δίκαιη και έχουμε εκατομμύρια θύματα και αδύναμα θεσμικά όργανα και μηχανισμούς. Ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι η δικαιοσύνη και τι χρειάζεται ε, έτσι ώστε τα θύματα να νιώσουν δικαιωμένα ε, και να επουλώσουν τις πληγές τους. και έχουν γίνει προσπάθειες ανακοχής ε, και συμφιλίωσης ε, διαφόρων τύπων διαδικασίες, μεταξύ αυτών και δικαστικές διαδικασίες, τα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε υπόψη όταν μιλάμε για τιμωρησία. Τρίτον, η <clears throat> ατιμορρησία ξεκινάει ώρες μετά τη διάπραξη ενός αδικήματος ατιμορρησία δεν σημαίνει ότι απέτυχε ένα δικαστήριο. Σημαίνει ότι απέτυχε η αστυνομία. Σημαίνει ότι ε, απέτυχε η έρευνα και η ανάκριση. Μιλάμε πολλές φορές για... Έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές ε, μια ακροματική διαδικασία που βρίσκεται στο τέλος της αλυσίδας, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε ένα πρόβλημα ατιμορρησίας πολύ πιο νωρί από όταν ξεκινούν οι αστυνομικές έρευνες. Έρευνες οι οποίες δεν συλλέγουν αρκετά στοιχεία, έρευνες που δεν παίρνουν καταθέσεις από τους κατάλληλους ανθρώπους, εξαιτία έλλειψη ικανοτήτων, έλλειψη πολιτική βούληση, εξαιτία πιέσεων ή φόβου. Οπότε η ατιμορρησία ξεκινάει από τη φάση της έρευνας και της ανάκρισης. Γι' αυτόν τον λόγο μία από τις συστάσεις μου στο πλαίσιο της ε, εργασίας μου για τον Τζαμάλ Κασόγκη είναι να δημιουργηθεί ένα μόνι, ένας μόνιμος μηχανισμός, διεθνής μηχανισμός για να εξασφαλίσει τις αμερόληπτες έρευνες. Αυτό θα είναι ένας μηχανισμός που θα αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και θα μπορεί να ξεκινήσει δικές του έρευνες, θα εντοπίζει την πιο κατάλληλη ε, δικαιοδοσία, εθνική ή διεθνή, για το κάθε αδίκημα. Μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, αν θέλετε, αργότερα. Πέμπτο σχολείο μου, νομίζω ότι είναι πέμπτο, λέει ο Μιλήτρια, το γεγονό ότι ένας από τους ε, πιο μεγάλους ενόχους ε, ε, διεθνώς που ε, ξεχνάμε πολύ συχνά είναι αυτοργή, ηθική αυτοργή. Ε, παρόλο ότι μπορούν να δικαστούν ως ε, ε, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών δεν εξασφαλίζουμε επαρκή διοξίτους. Όποτε μιλώ για τιμωρησία και για δικαιοσύνη, επιμένω στο ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε θεσμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να μπορούν να εργάζονται για αδικήματα από ένοπλες ομάδες και μη κρατικέ αρχές. Επίσης έχω να σας πω ότι έχω εργαστεί ε, σε διάφορα περιβάλλοντα για θέματα τιμωρησίας. Ο Τζαμάλ Κασόγγι ήταν μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες εργαστικά. Επίσης η σύγκρουση στο Ιράκ και αναζήτηση μιας προσωρινής δικαιοσύνης ή μάλλον ε, ε, ε, μιας ε, δικαιοσύνης μεταβατικής, καθώς επίσης ε, και την κατάσταση στη Μεσόγειο και στην Ιγυρία, που ήταν η τελευταία μου ε, επίσκεψη. Αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκα και μπορώ να σας σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ειρήνα. Ευχαριστώ πολύ. Σας επισκεφθήκαμε στην ε, αποστολή μας στη Νέα Υόρκη. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Που μας μιλάτε σήμερα για την ατιμορρησία. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένε περιπτώσεις, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα που υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το τελευταίο σας σχόλιο μου, θέλω να σας ρωτήσω, για, το, για την ατιμορρησία ε, θεσμών που δεν είναι κράτη, μη κρατικών θεσμών και κυρίως ενοπλών ομάδων. Συζητούσαμε για νωρίτερα εδώ ε, για πράξεις που λαμβάνουν χώρα από ομάδες ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις για παράδειγμα υποστηριζόμενες ενδεχομένως από το κράτος αλλά ίσως και όχι ε, αντικείμενα λοιπόν ε, με αυτούργο εταιρείε οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα μέσω δολοφονιών ανθρωποκτονιών είτε με πράξεις είτε με παραλήψεις όπως ε, για παράδειγμα ε, την καταστροφή του, πρόσφατη καταστροφή του φράγματος στην Βραζιλία. Ε, πώς μπορεί η διεθνής κοινότητα να διώξει πολυεθνικές συχνά εταιρείες που πολύ συχνά οι πράξεις τους διαπονται από ατιμορρησία. <laughs> Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγνες, για την παρουσίασή σου. Έχω ένα ερώτημα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά. Εσείς πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τη δουλειά που κάνετε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση που θέλετε σε διάφορες χώρες. Ας πούμε στις Φιλιππίνες είπατε ότι δεν είχατε πρόσβαση. Και για να μην στεναχωριέστε, ούτε εμεί μπορούμε να έχουμε πάντα πρόσβαση στι αποστολέ που κάνουμε. Οπότε για την πρόσβαση τι μπορούμε να κάνουμε και για τη χρηματοδότηση πώ μπορούμε να σα στηρίξουμε. Και επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση πού θέλετε να στηρίξει, σε ποιου άλλου τομεί θέλετε να στηρίξει τι προσπάθειέ σα. Για να το ζητήσουμε κι εμεί είτε από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλος κανείς. Εγώ θα είχα να κάνω μια ερώτηση, όπως και η Ειρήνα. Μιλήσαμε για την ευθύνη των ε, μεγάλων επιχειρήσεων ε, και το γεγονός ότι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως από τις συζητήσεις μας και τις συναντήσεις μας διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά υπάρχει μια συνενοχή ανάμεσα στα κράτη και τις πολυεθνικές. Έχουν κοινά συμφέροντα για παράδειγμα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, οι επιχειρήσεις ε, εκμεταλλεύονται ε, ανθρώπινους πόρους ή ορυκτά, αλλά έχουν άδεια από το κράτος και σε αυτή την περίπτωση αποσύουν τις ευθύνες τους. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ε, μου είπαν ότι η λύση δεν είναι απαραίτητα η δικαιοσύνη, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί κανόνες ε, ε, για τον σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των κοινωνικών και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να δώσουμε την εντύπωση στους πληθυσμούς που είναι υποεκμετάλλευση ότι πραγματικά εισακούνται. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε στους πολίτες την αίσθηση ότι πραγματικά τους σεβόμαστε και ότι μπορούμε να διώξουμε ή τα κράτη ή τις επιχειρήσεις που δεν ε, σέβονται τους πολίτες. you have the Ο Ε, είπατε ότι τα θύματα ε, νιώθουν απογοήτευση εξαιτία τη τιμωρησία. Όμω στην περίπτωση των ΗΠΑ Εθνών ε, πώ είναι το να μην είναι απογοητευμένα τα θύματα όταν στο Συμβούλιο ε, το Ανώτατο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν θέσει η Βενεζουέλα και η Κούβα. Και μάλιστα αμέσως μετά την έκθεση της είπα του ΟΗΕ που τις καταδικάζει. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ούτε εμείς. Έχετε το λόγο, Άγνες. Είναι ερώτηση ή δήλωση η δική σας, κύριε Λόπες. Uh, vote for uh, Ναι, ρώτησα για χώρε που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και παρόλα αυτά είναι μέλη του Συμβουλίου. Λοιπόν, για την εταιρική ευθύνη δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδική. και μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα στην εντολή μου δεν έχω επικεντρωθεί στο θέμα αυτό. Λίγο μόνο για την Ιγυρία και, την, ε, και τις Φιλιππίνες ε, ασχολήθηκα, οπότε θέλω να προσποιηθώ ότι έχω μια ειδική γνώμη να σας δώσω επί του θέματος. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας για τις ε, πολυεθνικές εταιρείε. Το πρώτο σημαντικό σημείο για μένα είναι να επιμείνουμε ότι το διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξελίσσεται μαζί με την εποχή. Ε, δημιουργήθηκε με βάση ένα σύστημα κρατών, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο διεθνές νομικό σύστημα που και γενικώ στη διεθνή κοινότητα που ζούμε πλέον, έχει, έχουν υπάρξει πάρα πολύ μεγάλες ε, περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων, ε, ιδιωτικοποιήσεων και της ασφάλειας. Μιλούμε και για ε, ιδιωτικούς ε, πολέμους πλέον. Το γεγονός ότι το νομικό σύστημα για τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα δεν δίνει νομική προσωπικότητα σε μη κρατικούς φορείς, όπως ας πούμε οι εταιρείε, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ναι, κάποια βήματα έχουν γίνει, κάποιε προσπάθειες έχουν γίνει. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα πριν από 25 χρόνια, μαζί με τον Άντριου Κλάπαμ, που είναι ειδικό για το θέμα. Σας ενθαρρύνω να τον προσκαλέσετε εδώ. Είναι πραγματικά ειδικό σε ό,τι αφορά την εταιρική ευθύνη. 25 χρόνια λοιπόν ξεκινήσαμε η πρόοδος ήταν να είναι πραγματικά πολύ μικρή. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα δόγματος και υπάρχει και πρόβλημα θεσμικό. Έχοντας ε, δουλέψει λίγο πάνω στα του δόγματος, έχω δει ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια, πολλοί δισταγμοί για να ζητηθεί διεθνής νομική προσωπικότητα για τις πολυεθνικές εταιρείε. Αν λοιπόν αυτό που θέλετε να κάνετε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε το δικό τους ρόλο ως παραβιαστές ας πούμε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσωπικότητά τους στο διεθνές, στη διεθνή σκακέρα. Αυτό δεν έχει γίνει. Ε, ούτε καλά ούτε ε, πλήρως. Και προφανώς αυτό έχει αντίκτυπο σε οποιοδήποτε δικαστικό σύστημα θέλετε να αναπτύξετε. Ας πούμε δεν μπορείτε να τους ε, θεωρήσετε υπόλογους στο δικαστήριο Μπορεί να τους θεωρήσετε ε, για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα. Μπορεί να τους θεωρήσετε υπόλογους για ε, παραβιάσεις ε, του εταιρικού δικαίου. Αλλά δεν θα θεωρηθούν υπόλογοι για την παραβίαση του δικαίου περί δικαιωμάτων. Και αυτό για μένα είναι πραγματικά ελλειπής ε, της πραγματικότητας και της εμπειρίας που έχουν τα θύματα των παραβιάσεων αυτών. Δεν έχω λοιπόν πιο συγκεκριμένη απάντηση να σας δώσω. Πέραν το ότι θα πω το εξή. Υπάρχει πρόοδος ως προς αυτή την πτυχή, δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο αρνητική, γιατί γίνεται και συζήτηση στη Γενέβη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχετική σύμβαση που βρίσκεται τώρα Υπάρχει λοιπόν αναγνώριση του φαινομένου και των ε, περιορισμών της νομοθεσίας για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα που βασίζεται μόνο στα όσα κάνουν τα κράτη και επίσης πρέπει οι, εταιρικοί, οι εταιρείες αυτές να ενταχθούν στο διεθνές νομικό ε, πλαίσιο που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία να εξηγήσει δημοσίως, να ε, εκδώσει δηλώσεις ότι υποστηρίζει, ας πούμε, την ε, ε, απόδοση νομικής προσωπικότητας στις πολυεθνικές εταιρείες για τα θέματα νομοθεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κάνει κάποια βήματα που θα μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η τελευταία συμφωνία για την συμφωνία για την ευθύνη συγγνώμη, των εταιριών ασφάλειας πάει λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, να ενισχύσει δηλαδή την αυτορυθμιστική βάση για την ευθύνη. Ακόμα όμως είναι ευθύνη του καθενός να το ρυθμίσει αυτό, της κάθε εταιρεία. Οποιαδήποτε προσπάθεια πάει προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω βέβαια εσείς πόσο, πόσο επιρροή μπορείτε να ασχίσετε, αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι, εταιρικές, οι εταιρείες να θεωρούνται υπόλογες για παραβίαση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελήφθη μια απόφαση πριν από 1,5 χρόνο περίπου που περιόρισε πολύ τη δυνατότητα να τους ε, θεωρήσουμε υπόλογους τους, ε, τις εταιρείες αυτές στα πλαίσια του Αμερικανικού δικαίου. Ε, οπότε έτσι ε, επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όμως ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που να έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν παραβιάσεις και εξωχωρικές και ενδοχωρικές αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε σε, εντός της ε, επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι εκεί φτάνει η εμπειρογνωμοσύνη μου για το θέμα αυτό. Και επίσης ε, εταιρείε είναι και το Facebook και άλλες τέτοιου είδους εταιρείες Οπότε η δική μου πρόταση είναι να μεταφερθούμε προς ένα σύστημα όπου αυτοί οι μεγάλοι παίχτες, πλατφόρμες επικοινωνίας, δεν ξέρω πώς τους λέμε ακριβώς, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται υπόλογοι σύμφωνα με μια διεθνή σύμβαση την οποία θα πρέπει και αυτοί να επικυρώσουν από κοινού με τα διάφορα κράτη. Δεν λέω ότι θα πρέπει να φτάσουμε ως εκεί πια, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουμε να να ρυθμίσουμε έναν κόσμο μέσα στον οποίο τόσες πολλές δραστηριότητες ιδιωτικοποιούνται. Και πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο ρόλος των ιδιωτικών εταιριών. Και στα πλαίσια πάντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εταιρείες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά Καλωσορίζουμε την βοήθειά σας στην προσπάθεια τη δική μας και στην ε, αποστολή. Ε, είναι αρκετά δύσκολη η εντολή που έχουμε. Πολλές χώρες ε, μας κρατούν τις πόρτες τους κλειστές. Εγώ πρόσφατα πήγα στην Ιγυρία και πραγματικά είμαι ευγνώμων στις Νιγηριανές αρχές που με κάλεσαν καταρχάς. Οπότε θα καλωσορίσω την βοήθειά σας και τη στήριξή σας. Και βεβαίως καλοδεχούμενη είναι και οποιαδήποτε δυνατότητα χρηματοδότησης για ειδικέ διαδικασίες. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, αλλά ο ειδικό εισηγητής εντός του συστήματος του ΟΗΕ δεν λαμβάνει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Υπάρχει βέβαια συνολικό πρόβλημα χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ σα μιλώ για το δικό μου πρόβλημα. Έχουμε ελάχιστη χρηματοδότηση. Πολλοί από του συναδέλφου μου δεν έχουν καν ε, στήριξη στη Γενέβη για την ε, δουλειά που κάνουν. Εγώ ευτυχώ έχω κάποια στήριξη, είμαι λίγο πιο τυχερή. Και πάντα είναι δύσκολο να κάνει κανείς κάτι. Ή τουλάχιστον για τη δική μου την ε, δουλειά. Είναι δύσκολο να γίνουν πράγματα χωρίς την ε, χρηματοδότηση. Η στρατηγική στήριξη βεβαίως είναι απαραίτητη. Αν δείτε δηλαδή όλα τα θέματα τα οποία με αφορούν και τα, με, τα οποία, με τα οποία ασχολούμαι είναι το, η παρακολούθηση της δολοφονίας του Τζαμαλ Κασόγγι, η ευθύνη των, για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στα πλαίσια του πολέμου Ιραξηρίας, ε, το ISIS, το Ισλαμικό κράτος, οι ξένοι μαχητές, το σύστημα που πρέπει να δημιουργηθεί και για την ε, δίκαιη δίκη και για την ε, απονομή ευθυνών. Για όλα αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί. Θα έπρεπε να είναι ένας από τους ε, μεγάλους ε, υπερασπιστές των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δική μου την οπτική, δεν ε, όσο δυνατά και ενεργά περιμέναμε. οι παραβιάσεις πάντα γινόντουσαν. Δεν είναι προϊόν του τελευταίου κύματος λαϊκισμού, υπάρχουν εδώ και καιρό. Η διαφορά αυτή τη στιγμή μεταξύ του τι αντιμετωπίζουμε τώρα και τι αντιμετωπίζαμε πριν 10 χρόνια είναι η σιωπή πολλών διεθνών φορέων. Είναι η σιωπή πολλών χωρών που θα έπρεπε και μπορούν να σταθούν απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις και να στηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν το κάνουν για λόγους που είναι πάρα πολύ βραχυπρόθεσμοι, πολύ κοντόφθαλμοι και δυστυχώς αποποιούνται και την ηθική που πτυχή και χρειά που δίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς αυτή είναι μια μάχη που χάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους παίκτες που λείπουν από τη διεθνή ε, σκακέρα. Και κάποια κράτη-μέλη. Στη δουλειά που έκανα για τον Τζαμάλ Κασόγγι, στην αρχή, αμέσως μετά τη δολοφονία του, υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες, πολύ στεναρές θέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους τελευταίους ε, τρεις-τέσσερις μήνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, θεσμικός φορέας και τα κρατη θέλουν να γυρίσουν σελίδα, να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό, δυστυχώς για κανέναν. Συμπεριλαμβανομένων και των Σαουδαράβων. Και είναι κρίμα. Η σιωπή, ας πούμε, για την κατάσταση στην Αίγυπτο είναι επίσης προβληματική. χρειάστηκε δυστυχώς να λάβω πολλές δηλώσεις ε, μαρτύρων για το τι γίνεται στην Αίγυπτο. Και η σιωπή γύρω από τις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εκοφαντική. Για το Ιράκ, η απουσία ηγεσίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, κυρίως ό,τι αφορά την ε, μετάβαση σε ένα ε, δικαστικό σύστημα μετά την στρατιωτική νίκη του Νοεμβρίου του 2017, ε, εκεί πληρώνουμε το τίμημα. Δεν υπάρχει στήριξη, δεν υπάρχουν επενδύσεις, ε, για την ε, επαναφορά της ασφάλειας στη χώρα, για την ε, δημιουργία δικαστικού συστήματος, για να υπάρξει ένα, μεταρρύθμιση των, του νομικού συστήματος. Εμείς επανειλημμένως έχουμε κατηγορήσει αυτές τις παράλογες δίκες που γίνονται τελευταίο 1,5 χρόνο στο Ιράκ. Και έχουμε Ευρωπαίους υπουργού που προσποιούνται ότι είναι κάτι σύνηθες οι δίκαιε ε, ξέρω ότι προσποιούνται, ξέρω ότι θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να το κάνουν και το ξέρουν και, αυτό, και αυτοί. Εγώ εκεί θέλω να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω στεναρέ δηλώσεις αρχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να επιβεβαιώσει τη σημασία των αξιών. Πέραν το να ε, ιδιωτικών των, των ίδιων συμφερόντων στρατηγικών ή πολιτικών. Θέλω ένα όραμα για την πολιτική διακυβέρνηση, για τη σταθερότητα και την ειρήνη και όχι κοντόφθαλμες ε, πρακτικές μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό θέλω να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος... Κούβα και Βενεζουέλα. Ναι, προφανώς είναι τραγική η κατάσταση. Κούβα, Βενεζουέλα, Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω και άλλες χώρες πώς εκλέγονται. Οι περισσότερες χώρες αυτές είναι μέλη περιφερειακών ε, ομάδων. Δεν εκλέγουν. Έχουν μια, ένα σύστημα κυλιόμενο, ας πούμε. Έτσι μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις. Έγινε μια προσπάθεια στις τελευταίες εκλογές Στην Κωνσταντίνα τώρα ήταν, δεν θυμάμαι, σε κάποια χώρα λατινοαμερικανική που υπήρξε μια προσπάθεια αποσταθεροποίηση του συστήματο που δεν ήταν επιτυχη. Η, αυτή λοιπόν η κυλιόμενη, αυτό το κυλιόμενο σύστημα είναι ένα σύστημα μυστικό προς το παρόν και έτσι φτάνουν εκεί που φτάνουν αυτές οι χώρες. Ευχαριστώ Άγνας. Δύο ακόμα ερωτήματα, η Ειρήνα και η Άννα. Ευχαριστώ. Ε, ένα ερώτημα για την Αίγυπτο. Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μελετά τα θέματα αυτά πολύ σοβαρά και τις χώρες αυτές, αλλά εμείς είμαστε μία επιτροπή μεταξύ πολλών και προσωπούμε ένα, ας πούμε, συμφέρον μεταξύ πολλών. Αλλά έχουμε αυξήσει την ευαισθητοποίηση προς αυτό και μπορώ με χαρά να σας πω ότι έχουμε Κάποιες μικρές επιτυχίες μεν, σημαντικές δε. Τον Οκτώβριο ο Ιμπραήμα Ζελντίν είχε εξαφανιστεί όταν α, αυθαίρετα συνελήφθη στις 11 Ιουνίου στο δρόμο και βρέθηκε ζωντανός, ακόμα βέβαια υπόκειται σε έρευνα, αλλά έχει επιβιώσει και είπε ο ίδιος ότι πιστεύει ότι αυτό έγινε λόγω της διεθνούς κατακραυγής που υπήρχε και όχι μόνο από την, την προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των ε, Επιτροπών ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Bundestag, στη Γερμανία. Εμείς είχαμε συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Γερμανικής Βουλής και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας για να ρίξουμε φως σε αυτές τις υποθέσεις. Και εγώ θα ήθελα να έχουμε πιο στενή συνεργασία με την κυρία Καλαμάρ και το γραφείο σας. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τις αναφέρουμε, να τις θίξουμε και στην Ολομέλεια, η οποία ούτως ή άλλως γίνεται κάθε μήνα. Ευχαριστώ. Η Άννα εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ακριβή απάντησή σα για το τι θα πρέπει ή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω κι εγώ να επαναλάβω αυτό που είπε η Ειρήνα. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φυσικά υποστηρίζουμε πλήρως τους ε, σκοπούς ε, που έχετε και ξέρουμε η ειρηνα Εμεί εδω στην επιτροπη ανθρωπινων δικαιωματων χρειάζεται και στήριξη και χρηματοδότηση. Οπότε εγώ θα σα ενθάρρυνα να είσαστε σε επαφή μαζί μα αν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα ή αν βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να σα βοηθήσει να δουλέψετε καλύτερα και εμεί να χρησιμοποιήσουμε όποια όπλα έχουμε, ώστε να πιέσουμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία ενιαία ε, προσωπικότητα, είναι πολύ, ε, έχει πολλά πρόσωπα. Και επίσης να πω ότι συμμερίζομαι τα όσα είπατε για το Ιράκ. Αν δούμε την κατάσταση στο Ιράκ τώρα, φαίνεται ότι τα προβλήματα υπάρχουν και δεν έχουμε βρει τελικώ ε, διαδικασίες για μετάβαση σε ένα ε, σόφρον δικαστικό σύστημα. Βεβαίω, ε, προφανώ είναι δύσκολο αυτό μετά από τέτοιε ακραίε επιθέσει. Μιλήσατε και για τον Άισι, για το Ισλαμικό κράτο. Ε, κάτι για το Ιράκ και τη Συρία που αναφέρατε. Έχουμε περίπου 70 ε, Μαχητέ του ε, ε, Ισλαμικού κράτου σε στρατόπεδα. Το Ιράκ έχει ξεκινήσει δίκες και τις, τους εκτελεί. ήδη 20.000, 2.000 συγγνώμη, έχουν εκτελεστεί, αλλά η δική σας, το δικό σας σκεπτικό ποιο είναι, τι τι κάνουμε με αυτούς τους 70.000 που είναι στα, στα στρατόπεδα. Υπάρχουν και κάποιες ιδέες για δικαστήρια ad hoc. Ε, δεν έχω βέβαια καλύτερη άποψη για αυτά, αλλά δεν έχω και καλύτερη επιλογή. Επίσης, τα ρομπότ που δολοφονούν ε, τα έχετε υπόψη, έχετε, ε, έχετε ασχοληθεί με την παρέμβασή τους με τα ένοπλα ντρόν και τα ρομπότ. Ε, γιατί και αυτά ε, εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εξοδικαστικές δολοφονίες. Και εκεί μπορεί να υπάρχει το θέμα της ατιμορρησίας. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω δύο ερωτήσεις συχνά έχουμε ακτιβιστές που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δολοφονούνται τελικά, ηγέτες που δολοφονούνται. Και συχνά πίσω από αυτά τα εγκλήματα, αν δεν μπορούμε να βρούμε ποια είναι η ευθύνη του κράτους, ε, βρίσκουμε εγκληματικές οργανώσεις που τα κράτη ε, θεωρούν ότι όλα αυτά είναι διευθέτηση λογαριασμών μεταξύ συμμοριών, έχουν σχέση με τον αρκεμπόριο όπως στην Κολομβία κτλ. Ενώ στην ουσία πρόκειται για δολοφονίες ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε ε, συμπεριλάβει αυτές τις ενώσεις μέσα σε αυτά τα non-state actors, τα οποία αναφέρεται τους μη κρατικού παράγοντες και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση για να πατάξουμε την ατιμορρησία που σχετίζεται εδώ με το κράτος. Επίσης, το πλαίσιο πλαίσιο της αποστολής σας. Ε, έχετε εξετάσει ευρωπαϊκές περιπτώσεις. Έχουμε τρεις περιπτώσεις δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν στην Ευρώπη και που έχουν προφανείς ε, σχέσεις με διερεύνηση γύρω από υποθέσεις διαφθοράς ή ατασταλίες βάρος του κρατικού χρήματος. Έχουμε δημοσιογράφους, δημοσιογράφο από τη Σλοβακία, έναν από τη Βουλγαρία και έναν από τη Μάλτα. Μπορείτε να διερευνήσετε τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, το κάνατε και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω από την τελευταία σας ερώτηση όσον αφορά αυτούς τους τρεις Ευρωπαίους δημοσιογράφους. Ο συνάδελφός μου David Cake είναι ο ειδικό ε, εισηγητής για την ελευθερία της έκφρασης ε, και ε, σε μια δημόσια ανακοίνωση επίσης αποφανθήκαμε για την δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Καρουάνα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από αυτά που έγιναν λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες και που έδειξαν κατά τη γνώμη μου ότι η επιμονή και η αποφασιστικότητα της κοινωνίας των πολιτών μπορούν τελικά ακόμα να, κάνουν, να κινηθούν ακόμα και οι ε, πιο ε, διστακτικές ε, κυβερνήσεις, αυτές που δεν θέλουν να κινητοποιηθούν. Ο Πρωθυπουργό της Μάλτας ανακοίνωσε την παρέτησή του ε, τον ερχόμενο Ιανουάριο και αυτός που έδωσε την παραγγελία του φόνου ταυτοποιήθηκε τελικά. Σε αυτή την ανακοίνωση λοιπόν, σε αυτό το ανακοινωθέν τύπου που ε, βγάλαμε σήμερα, ζητάμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή Δημόσιας Έρευνας που συστάθηκε μετά την ε, έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, και του εισηγητή, δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του, Πίτερ, Πίτερ Χόμστ, νομίζω λέγεται, ζητήθηκε λοιπόν να συσταθεί μια επιτροπή εγκρίθηκε η σύστασή της και θα αναλάβει εργασίες στις 6 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα για αυτή την σύσταση και ζητάμε η Επιτροπή να μπορέσει με αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο να εργαστεί. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση ε, συμφερόντων και σε καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργό δεν θα παίξει οποιοδήποτε ρόλο στο έργο αυτής της Επιτροπής. Αποτελείται από τρεις επιφανείς νομικούς, τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα και για μας αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Όπως βεβαίως είναι και η έρευνα η αστυνομική ε, που έλαβε χώρα αυτές τις τελευταίες μέρες. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσφέρθηκα να συναντήσω την ε, Επιτροπή που έχει αναλάβει την έρευνα και βεβαίως μπορώ να, σας τους ενημερώσω για την έρευνά μου για τον Τζαμέλ Κασόγγι. Γιατί αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν διαβάζουμε τους όρους, ε, πρόκειται για δίκαιο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποινικό δίκαιο μαζί. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εγώ έκανα τη δική μου έρευνα για τον Τζαμάλ Κασόγγι, η δική μου έρευνα βασιζόταν κυρίως στο ανθρωπιστικό δίκαιο και το ε, διεθνές δίκαιο. Ε, πήγα λίγο παραπάνω στα χωράφια του ποινικού δικαίου, αλλά δεν είναι αυτή η αποστολή των ειδικών ε, εισηγητών. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω ε, μια παρακολούθηση με βάση το ποινικό δίκαιο περισσότερο παρά το ανθρώπινο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τα δύο δίκαια βεβαίως είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει να αποδοθεί, να προσδιοριστεί η ευθύνη του κράτους και η μεμονωμένη ποινική ευθύνη. Γιατί και τα δύο μετράνε. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με αυτούς τους όρους, με τα κριτήρια αναφοράς και βεβαίως θα παρέχω ε, στήριξη όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τα έργα. Αυτά για την δημοσιογράφο. Όσον αφορά τώρα την ε, μεταβατική δικαιοσύνη στο Ιράκ. Στεναγμός. Από πού να αρχίσουμε. Είναι πολύ δύσκολο όταν σκέφτεται κανείς ε, την κατάσταση να μην ε, έχει μια μικρή πικρία για όλα αυτά τα χρόνια που κατασπαταλήθηκαν. Και θέλω να εκφράσω αυτή την πικρία για λίγο. Μετά το 2017 η κυβέρνηση του Ιράκ έκανε συλλογικές ε, δίκες και βεβαίως πολύ γρήγορα ε, καταγγέλθηκε ότι δεν ήταν δίκαιες δίκες. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα, θα ήταν επίγον να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, να πιέσουμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, το Ιράκ για να κάνει μια μεταρρύθμιση ε, των, ε, του δικαστικού του κλάδου και των δικών. Διαφορετικά δεν ε, θα υπάρχει, δεν μπορούμε να ε, τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους ε, των ε, φρικτών ε, γεγονότων. Το θέμα δεν είναι να αποδώσουμε δικαιοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει η δικαιοσύνη, η απονομή της δικαιοσύνης, όχι μόνο για να τιμωρηθούν οι δράστες που ε, για μένα ίσως είναι το λιγότερο, αλλά κυρίως για να δικαιωθούν τα θύματα. Οι φρικαλιότητες που έχουν γίνει από το ΆΕΣΙΣ και από όλους όχι μόνο εδώ παραβιάζεται η δίκαιη δίκη, αλλά παραβιάζονται τα ίδια τα δικαιώματα των θυμάτων θυμάτων που δεν μπορούν να παραστούν. Δεν έχουν διερευνηθεί υποθέσεις τα θύματα του ISIS πηγαίνουν στην αστυνομία και τέρμα. Μετά δεν υπάρχει καμία παρακολούθηση. Μιλάμε για ατιμορρησία. Και εδώ έχουμε θύματα που δεν εισακούονται καν, όχι να πηγαίνουν τελικά ε, να δικάζονται οι υποθέσεις τους. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με, δίκες αστραπή, όπου δεν δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες. Και εγώ εργάστηκα ε, σε ε, περιπτώσεις πέντε ηγετών του ΆΕΣΙ, σε πολύ ψηλό επίπεδο δηλαδή, πριν από κάποιους μήνες. Έγιναν οι δίκες πριν από 8 μήνες. Η δίκη αυτή πέρασε εντελώ απαρατήρητη από τη διεθνή κοινότητα και τουλάχιστον ένα από αυτά τα άτομα δημοσία αποδέχτηκε ότι ήταν ένοχος εγκλημάτων πολέμου στη Μοσούλη. Ποιο το ξέρει όμως, κανένας. Μίλησα με Σύριους που αγαπημένοι τους είχαν εξαφανιστεί, τους είχε απάγει το και χιλιάδες, όπως και χιλιάδες άτομα και που ίσως βρίσκονται σε ομαδικούς τάφους και μου είπαν δεν θα ανοίξουμε αυτούς τους ομαδικούς τάφους γιατί υπάρχουν ακόμα άτομα στις ε, φυλακές του Ιράκ που μπορούν να μας πούν πού σκοτώθηκαν τα οικοί μας και πού βρίσκονται. Αυτό θα είναι το λογικό βήμα, αυτή είναι η λογική έρευνα, η οποία όμως δεν έχει γίνει. Λυπάμαι που σας τα λέω όλα αυτά και φαίνομαι τόσο απογοητευμένη. Ναι, είμαστε μία διεθνής ομάδα. Έχουμε συλλέξει στοιχεία αποδεικτικά και μπορέσαμε έναν στους 28 ηγέτες του ISIS να τον δικάσουμε. Είναι μια αρχή. Σίγουρα είμαι υπέρ αυτού, σίγουρα χαιρετίζω το γεγονός και ελπίζω ότι τελικά η δίκη, οι δίκες αυτές, θα είναι μια ευκαιρία απονομής δικαιοσύνης για μας και τους Ιρακινούς. Αλλά η δική μας ευθύνη τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό με ενοχλεί εμένα προσωπικά, ακριβώς είναι το μερίδιο ευθύνης που φέρουμε. Ναι, είναι πολύπλοκες αυτές οι δίκες να συσταθούν αυτά τα δικαστήρια, αλλά η στήριξη της κυβέρνησης του Ιράκ για μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος σίγουρα δεν είναι εύκολο. Τους έχω συναντήσει, έχουμε συζητήσει για τη μεταβατική δικαιοσύνη, πολλά τα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά αυτό πρέπει να γίνει. Βεβαίως γνωρίζετε την κατάσταση, όπως και εγώ. Και όσον αφορά τώρα τους ξένους μαχητές, Αναμφισβήτητα, για μένα, δεδομένη της σημερινή κατάστασης, η μόνη εναλλακτική είναι να επιστρέψουν για να δικαστούν. Αυτό θα επιτρέψει μια συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ ανθρώπων που έχουν αποδεικτικά στοιχεία, που έχουν συλλέξει τα τελευταία χρόνια και να γίνει λοιπόν κάτι που να καταλήξει σε μία δίκη. Και μια που μιλάμε για τιμωρησία, να σας πω και το εξή. Εάν ένας στρατηγός, για παράδειγμα, του Συριακού στρατού, πάει στη Γερμανία ως πρόσφυγας και ταυτοποιηθεί, θα δικαστεί και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες ε, που έχουν να κάνουν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν όμως κάποιος από το ISIS, ε, υψηλά ιστάμενος, βρισκόταν στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, θα δικαζόταν ε, σύμφωνα με τον εγχώριο αντιτρομοκρατικό νόμο, όχι με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Γιατί χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο καθεστώς κατά της ε, τρομοκρατίας και σε, ε, όπως για τον ISIS για παράδειγμα, και τελικά ε, δίνουμε πολύ λίγα περιθώρια στα θύματα. Στη Γαλλία έγιναν κάποιες δίκες που είχαν ως επίκεντρο τα θύματα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν φτάνουμε σε μια δίκη επί τη βάση του αντιτρομοκρατικού νόμου, ε, τα θύματα δεν μπορούν να καταθέσουν και δεν παρίστανται. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα στο Ιράκ ε, και για τους ε, ηγέτες του ISIS ότι δικάζονται όχι για τους βιασμούς, όχι για την καταναγκαστική δουλεία, όχι για τις, α, τους μαζικούς φόνους, αλλά ως, αντιτρομοκρατική, ως, τρομοκρατική οργάνωση. Όταν λοιπόν μιλάμε για ε, τιμωρησία, ναι, μπορεί να τους καταδικάζουν τελικά σε θάνατο, σύμφωνα με το νόμο του Ιάκ, αλλά δεν έχει αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη, δεν είναι δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Συνεργάζομαι λοιπόν με παραγόντες στο Ιράκ ε, για να βρούμε ποια θα είναι η πιθανή συνέχεια. Συναντάω, ε, θα συναντήσω σε λίγες μέρες μέλη οργανώσεων πολιτών για να καταλάβουμε, να καταλάβουμε καλύτερα τη σκοπιά των θυμάτων και όχι τη σκοπιά του κράτους. Για να δούμε πώς οι ίδιοι επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη από τη δική του σκοπιά. Θα είμαι εκεί σε λίγες μέρες. Όχι, δεν θα μιλήσω για τους ε, διαδηλωτές. Όχι, αυτό δεν το θίγω. Και για την ενημέρωσή σας, ήμουν στο Ιράκ ε, πριν από δύο χρόνια περίπου και συνάντησα τον υπεύθυνο για τους μαζικούς τάφους. Ήταν τον Νοέμβριο του 2017 και υπήρχαν κάποιοι μαζικοί τάφοι που είχαν σχέση ε, με τον Άισις κατά τελευταία γεγονότα και μου είπαν ότι θα χρειάζονταν 800 χρόνια με βάση τους πόρους που διαθέτουν σήμερα για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. και δεν μιλούσαν για τους ε, τάφους που υπήρχαν ήδη από πριν, τους μαζικούς, ε, λόγω της ε, εισβολής της Αμερικής ή όπως θέλετε πείτε την. Έχουν βρεθεί έκτοτε πολύ περισσότεροι μαζικοί τάφοι. Αυτό σας δίνει λοιπόν μια ιδέα του τι συμβαίνει και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας ως διεθνή ε, κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια ε, πολεμάμε ε, μια οργάνωση που έχει πραγματικά διαπράξει φρικαλαιότητες και σήμερα, τη στιγμή που μπορούμε να απαιτήσουμε να δοθεί δικαιοσύνη, τελικά δεν υπάρχει κανένας, τίποτα. Κανένας που να μπορεί για αυτή την περιοχή του κόσμου να εκφράσει ένα όραμα μεταπολεμικό. Και αυτό πραγματικά ε, είναι τραγικό. Moving on. Συνεχίζουμε. Οι εγκληματικέ οργανώσει, καρτέλ, συμμορίε και τέτοια. Χαίρομαι που θέσατε αυτό το, την ερώτηση, αλλά δεν έχω απάντηση. Είναι τμήμα της δικής μου διαδρομής ως αγωνιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων την δική μας δουλειά προτείνουμε ε, να κλείνουμε τα μάτια, να ξεχνάμε μάλλον ε, τις ε, που διαπράττουν εγκληματικές οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας ε, με τους καθημερινούς ανθρώπους, είναι τα, πιο, τα, τα πρώτα βία επεισόδια τα οποία τα οποία καταγγέλουν. Και έχω μάθει πλέον να μην αγνώ τέτοιου τύπου βίες πράξεις που δεν καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω εργαστεί με συμμορίες σε μία αποστολή στο Ελσαλβαδόρ. Εστίασα και στις παραβιάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και στις παραβιάσεις εκ μέρους των συμμοριών. Το σημείο αφιτερίας μου είναι ότι αυτές οι συμμορίες, στο Μεξικό μπορεί να είναι και καρτέλ μάλιστα, ελέγχουν συγκεκριμένες περιοχές, ελέγχουν ανθρώπους, ελέγχουν όργανα του κράτους, κρατικά όργανα, παρόλο που τα κράτη πολλές φορές δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Οπότε εξαιτία αυτού του ελέγχου εξαιτία του γεγονότος ότι κατά κάποιο τρόπο ασκούν κυβερνητικές αρμοδιότητες. Το Ελσαρβαδόρ, για παράδειγμα, υπάρχουν συμμορίες οι οποίες παίζουν ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Ε, σε άλλες περιοχές ε, εισπράττουν φόρους, δίνουν δάνεια. Εξαιτία αυτού, εξαιτία του γεγονότος ότι οι συμμορίες μερικές φορές υποκαθιστούν κρατικές λειτουργίες, υποκαθιστούν το κράτος. Ε, το κράτος λοιπόν δεν χάνει απλώς τη μάχη στρατιωτική, αλλά χάνει και την πολιτική μάχη μερικές φορές. Χρειάζεται λοιπόν εξαιτία αυτού να αλλάξουμε νοοτροπία μερικές φορές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσφατα ε, ανακοίνωσε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία εναντίον το καρτέλ του Μεξικού. Το ανακοίνωσε μετά την πρόσφατη δολοφονία ε, ε, μεξικανοαμερικανικών οικογενειών μαζί με τα παιδιά τους. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό. Είναι αναποτελεσματικό όμως όπως είναι αναποτελεσματική και οποιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση εναντίον ομάδων οι οποίες δεν είναι απλώς βίες αλλά ασκούν και κυβερνητικές εξουσίες. Η φύση του κοινωνικού συμβολέου μεταξύ αυτών και της κοινωνίας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε αυτό το θέμα το ζήτημα των συμμοριών, γιατί αλλιώ δεν θα βρούμε λύση. Δεν έχω λύση. Στην έκθεσή μου λέω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα πραγματικά το σύστημα διακυβέρνηση αυτών των ομάδων. Διότι δεν λειτουργούν μόνο μέσω της βία, παρόλο που η βία συχνά είναι μεγάλο κομμάτι της δράσης τους συχνά οι δράσεις τους ε, έχουν ε, ιστορικό υπόβαθρο ή έχουν ένα υπόβαθρο ε, συγκεκριμένων παραπώνων τη μεριά του λαού. 20 χρόνια σκληρής και ανελαιού στρατιωτικής κατασταλτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των συμμορίων στη Λατινική Αμερική δεν έδωσαν τίποτα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, υπόδειγμα. Δεν βλέπω κάποιο άλλο τρόπο. Euh, euh, Ευχαριστούμε, Αγνές. Πολύ εντυπωσιακά όσα μας είπες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι, οι εκθέσεις σας, οι εισηγήσεις σας στο πλαίσιο της ε, δουλειάς σας ε, ε, στον ΟΗΕ, στην Επιτροπή ΔΕΒΕ μιλήσαμε για τη σύνδεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτοπισμένων ανθρώπων δουλειά που γίνεται στον ΟΗΕ και νομίζω ότι και η δική σας δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική. και θα μας έχετε δίπλα σας για να μεγενθύνουμε και να διαδώσουμε το μήνυμά σας. Θα είμαστε η ηχό της δουλειάς σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω, το λόγο, θα δώσω την προεδρία στην Ειρήνα για να δούμε το επόμενο σημείο που έχει σχέση με την Αίγυπτο. Oui. Και κλεισμένο των θυρών. L'échange de vue sera in camera.